από τις Λιβικές αρχές στον χώρο της, της ασφαλείας και της δημοκρατίας για τη μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Έχω έξι προτάσεις ψηφίσματος που θα ψηφιστούν μετά τη λήξη της συζήτησης. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία ως ήθιστε, θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Οπότε σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. je hlasování o Θα ψηφίσουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ιδιαίτερα όσον αφορά το θάνατο του blogger Σατάρ Μπεχέστη. Επτά πολιτικές ομάδες έχουν υποβάλει τις προτάσεις αυτές ψηφίσματος. Και έχουμε και ένα νέο κείμενο. Δεν βλέπω να έχετε παρατηρήσεις. Συνεπώς ψηφίζουμε. Παράγραφος 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Η ε, κυρία Ντεκάισερ. Παρακαλώ, κύριε Ντεκάισερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τεχνική βέβαια η τροπολογία αυτή, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το κείμενο, με τη διατύπωση. Ο κύριος Παναγή Ζαφάρ νομίζαμε ότι ήταν στη φυλακή ακόμα, οπότε το τροποποίησαμε. Είναι ε, ελευθερωθεί. Είναι στη διαδικασία της έφεσης, αλλά έχει ελευθερωθεί. Οπότε πρέπει να αλλάξει ο χρόνος, <clears throat> να μην πούμε ότι is serving jail, αλλά was και μετά να λέμε ότι ο Ζαφάρ Παναγί κάνει έφεση για έξι χρόνια φυλακή και για το πάγωμα, για την ποινή που το επιβάλλανε και για το πάγωμα των λογαριασμών του. Ενώ η, το άλλο βραβείο Ζαχάροφ είναι σε απεργία πείνας. Ευχαριστούμε. Λέω πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνατε. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρώτας ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. εγκρίνατε. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, όσον αφορά τις ψηφοφορίες πάντα. Και αυτή είναι η ψηφοφορία που έχουμε με έξι προτάσεις ψηφίσματος για την κατάσταση στη Βυρμανία. Ιδιαίτερα για τις συνεχιζόμενες ε, διότητες στην πολιτεία Ρακίτ. Κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων. Δεν υπάρχουν ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, ψηφίζουμε τώρα έξι προτάσεις ψηφίσματος όσον αφορά την κατάσταση των μεταναστών στην Λιβύη. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Καλησπέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες για σήμερα. Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περίοδου συνόδου. Αν δεν υπάρχουν ε, σχόλια, επί των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν σήμερα θα απευθυνθούν